είναι με δυόμιση και τρεις, η ώρα με έντεκα. Μπορείτε να βρείτε στο website του Κοινοβουλίου την ημερησία διάταξη. Πέρα στη συνεδρία σας.